εξηγήσει ψήφου. Παρακαλώ όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να το κάνουν ήσυχα. Για να ακούσουμε τις επεξηγήσεις επί των κειμένων που ψηφίσαμε σήμερα. Παρακαλώ συνάδελφοι ε, αποχωρήστε ησύχω ε, για να μπορέσουν όσοι θέλουν να λάβουν το λόγο να μιλήσουν ήσυχα και να ακουστούν επεξηγήσει ψήφου επί των σημείων που ψηφίσαμε σήμερα. Σας ενημερώνω ότι έχουμε πάρα πολλού που έχουν δηλωθεί για να ε, κάνουν επεξήγηση ψήφου, αιτιολόγηση ψήφου. Μέχρι τις 3 παρατέταρτο μπορούμε να συνεχίσουμε. Ε, χρειάζεται χρόνος για προετοιμασία της αίθουσας ε, για να συνεχίσουμε στις 3. Οι επόμενες αιτιολογήσεις θα ε, δοθούν αύριο ε, και ε, οι υπόλοιπε μπορούν να υποβληθούν γραπτός. Παρακαλώ, περάστε έξω από την αίθουσα για να συζητήσετε, για να λάβουν τον λόγο οι συνάδελφοι για την αιτιολόγηση ψήφου. Ε, αποχωρήστε από την αίθουσα ήσυχα. Ο κύριος Πέτερ Γιάρ έχει το λόγο για ένα λεπτό για την έκθεση Ζωάου Φερέρα, Συμφωνία Αλληλευτικής Σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου, Αλληλευτικές Δυνατότητες και Χρηματική Αντιπαροχή, ο κύριος Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε. Ένα λεπτό. Θα ήθελα να μιλήσω για όλες τις ε, συμφωνίες αλληλευτικής σύμπραξης. Ε, ε, βεβαίως μιλάμε για win-win καταστάσεις, έχουμε συμπράξεις και δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, όμως θα ήθελα να παρακαλέσω η αρμόδια επιτροπή να κάνει και εκ των, έλεγχο και να μην χαλαρώσει διότι πρέπει να δούμε αν υπάρχει υπεραλίευση πέρα από τις δυνατότητες και επίσης πρέπει να εξετάσουμε ενδελεχώς τα κονδύλια που καταβάλλονται ε, αν όντω αυτά ε, χρησιμοποιούνται για αναπτυξιακά προγράμματα και δεν ε, κολλάνε στη διοίκηση. Ε, υπ' αυτές τις προϋποθέσεις συμφωνώ και ελπίζω ότι εκ των υστέρων έλεγχος και προετοιμασία θα, θα γίνει σωστά στην αρμόδια Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζόναθαν ε, για την ε, ε, έκθεση για τη Μαδαγασκάρη. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Θεωρώ, κυρία Πρόεδρε, ότι οι συμπράξεις αυτές χαρακτηρίζονται από ένα κοινό στοιχείο ότι δηλαδή δίνουμε χρήματα σε πολύ φτωχέ χώρε, ώστε να μας αφήσουν να καταλυστεύουμε τους φυσικούς πόρους τους. Ιδιαίτερα η Μαδαγασκάρη έχει μια ιδιαίτερη οικολογία, χλωρίδα και πανίδα πολύ ε, ποικιλόμορφη σε ό,τι αφορά ε, σε σχέση με τις διαφορετικές περιοχές. Χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία, ειδική μεταχείριση και δεν νομίζω ότι αυτή η συμφωνία κατά ανάγκη καλύπτει τις ανάγκες της Μαδαγασκάρης. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η έκθεση Σκά Κέλλερ ε, για τα μέτρα υπέρ της Ιταλίας και Ελλάδας ε, προσωρινά μέτρα στο τομέα της διεθνούς προστασίας. Ε, ε, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί δεν ψήφισα υπέρ της έκθεσης Κέλλερ. Όχι γιατί δεν συμφωνώ με την ελληνική. Το αντίθετο μάλιστα είναι απαραίτητη και δείχνει ανθρωπιά. Αλλά θα ήθελα ε, να δοθεί βοήθεια ε, και στις, στις οικογένειες χριστιανών που φτάνουν στην Τσεχία ε, καταδιακόμενοι από τα Ισλαμικά κράτη. νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε υπάρξει συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των χωρών για την κατανομή των 40.000 προσφύγων. Αυτό είναι ένα απαραίτητο σημείο αυτού του θέματος ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν οι υπεύθυνοι της ε, πολιτικής ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι να παίρνει αποφάσεις η Ελεονόρα Φροέντσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ στήριξα την έκθεση Κέλλερ γιατί με έπεισε, ε, γιατί πιστεύω λοιπόν ότι ε, είναι, ε, λαμβάνει υπόψη ε, σημαντικό σημείο ε, οι 40.000 πρόσφυγες να αφορούν μία πρώτη φάση και να αποτελέσουν μία αρχή που θα ακολουθηθεί και από άλλους πρόσφυγες. Ε, πιστεύω ότι καθόλου δεν αρκούν αυτά που ακούσαμε το πρωί από τον πρόεδρο Γιούγκερ και νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν διαρκώς να γίνεται η διαφοροποίηση ανάμεσα σε οικονομικούς μετανάστες και πρόσφυγες. Νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται για να προστατευτεί ε, ε, το δικαίωμα στο άσυλο, αλλά ε, για άλλους λόγους. Θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία όσον αφορά το άσυλο. Θα πρέπει να γίνει πιο η χώρα υποδοχής η Ευρώπη και να αλλάξει το Δουβλίνο. Ευχαριστώ. Κέρζη, πώς πισήλε ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ψήφισα υπέρ της προσώστοσης που αναφέρεται στην έκθεση. Είμαι πεπισμένος ότι στην πράξη όμως αυτό δεν θα λειτουργήσει ο σύστημα. Πιστεύω ότι οι αιτούντες άσυλο πρέπει να ζητήσουν άσυλο όπου επιθυμούν να εγκατασταθούν. Εκείνο το κράτος μέλος πρέπει να λάβει την απόφαση, εφόσον βεβαίως πληρούνται οι διεθνείς προϋποθέσεις και όροι. Νομίζω ότι το μέτρο είναι λάθος, ε, είναι κατά των συμφερόντων των ετούντων άσυλο και δεν θα λειτουργήσει στην πράξη το σύστημα. Ούτως ή άλλως θα πάνε εκεί που θέλουν, εκεί που είναι οι οικογένειές τους. Και σε τελευταία ανάλυση αυτή η διοικητική ανακατανομή των ετούντων άσυλο ε, οδηγεί ουσιαστικά σε ε, καταστάσεις ε, ε, ο χείρος της Ευρώπης είμαι υπέρ της αλληλεγγύης όπως η τσεχική κυβέρνηση αλλά κατά της ανακατανομής μέσω διοικητικών μέτρων. Η κυρία Νίνα Τζιλ. Γκίλ. Εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο... Εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο ε δείξαμε ε, την αλληλεγγύη μας ε, και ανέκαθεν και μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο ε, δείξαμε την αλληλεγγύη μας απέναντι σε όσους έφευγαν από εμπόλεμες περιοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους πρόσφυγες από την Συρία Υπάρχουν 3.000 ασυνόδευτα παιδιά στους καταβλισμούς στην Ιταλία. Τι γίνεται για να φροντίσουμε ότι μονίμως ε, θα ε, κατανεμηθούν σε κάποια χώρα και θα προστατευθούν και θα υποστηριχθούν. Ε, είναι σαφές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και θα πρέπει αυτό να το κάνουμε τώρα. Γι' αυτό είμαι υπέρ της έκθεσης Κέλλερ. Ευχαριστώ κυρία Γκίλ. Επόμενος μιλητής ο κύριος Στάνισλαφ Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να πω ότι ήμουν υπέρ της έκθεσης Κέλλερ. Δεν, ωστόσο, ε, δεν είμαι υπέρ του, της υποχρεωτικής ποσόστοσης και σας εξηγώ, ε, αναφέρεται στη βίβλο ότι δεν υπάρχει πίστη χωρίς δράση και πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μιλήσουμε ε, για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε στο όνομα αυτής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης την Ιταλία και την Ελλάδα. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει με τις ποσοστώσεις, αλλά ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει κατά αυτή την έννοια μια συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών. Χωρίς αλληλεγγύη δεν είναι δυνατόν δυνατόν ε, να πει κανείς ότι έχει πίστη στην Ευρώπη ή πίστη ε, γενικά. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κυρία Κριστίνα Μορβάη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Φυσικά, εγώ ε, καταψήφισα την έκθεση αυτή, αλίμονο. Και είχε τη γνωστή κατάληξη και αυτή η συζήτηση. Δεν απαντήθηκαν οι ερωτήσεις μας. Μας είπαν ότι θα πρέπει η Ουγγαρία να τηρεί το Σέγγεν, ε, τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα. Ε, ε, και κοινοτοπίες ακούσαμε ότι τόσοι μετανάστες και τόσοι πρόσφυγες θα πρέπει να γίνουν δεκτοί με διάφορους λόγους και δικαιολογίες. Εύκολο είναι να το λέει κανείς αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. δική του ζωή και η δική σας δεν πρόκειται να αλλάξει σίγουρα, ανεξαρτήτως του αριθμού των προσφύγων. Ε, θα έρχεται να σας παίρνει η μαύρη σας Mercedes, θα μένετε σε πολυτελή ξενοδοχεία, δεν θα μειωθεί ο μισθός σας, μένετε σε ωραίες πολυτελείς συνοικίες κτλ. Ποιος ζει στην ίδια συνοικία με τους πρόσφυγες και τα παιδιά σας έχουν εύκολη ζωή και ε, όταν ε, δεν θέλετε να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους μετανάστες, τα βάζετε σε ιδιωτικά σχολεία, σε ιδιωτικά νοσοκομεία και είστε μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τζαμπάνσκι, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μιλάμε για δεσμευτικές ποσοστώσεις για τους πρόσφυγες. Ε, είμαι κατά, γιατί αυτό είναι κατά της, κυριαρχικής, της κυριαρχίας των κρατών μελών, που πρέπει να μπορούν να ελέγχουν τα σύνορά τους. Είμαι κατά Επίσης, διότι το επίπεδο διαβίωσης στα κράτη-μέλη είναι διαφορετικό. Πώς μπορείς να βάλεις τον κόσμο να μείνουν στην ε, Ουγγαρία, τη Γερμανία ή τη Σουηδία. Ε, ε δημιουργούνται διακρίσεις ε, μεταξύ των προσφύγων. Επίσης, ποιος είναι ο πρόσφυγας και ποιος είναι ο παράτυπος μετανάστης. Δεν είναι σαφής η διαφορά. Δεν... Ε, είναι πλήρης ο ορισμός, ούτε υπάρχει σαφήνεια πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε παράλληλα δεσμευτικές ποσοστώσεις, διότι θα πρέπει να φιλοξενήσουμε στο τέλος εκατοντάδες εκατομμύρια. Η Συμφωνία Σέγγεν επίσης απεδείχθη αναποτελεσματική όπως και ο κανονισμός ε, του Δουβλίνου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έθερδιτζε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μιλάμε για μέτρα που ανοίγουν διάπλατα τις πύλες της Ευρώπης για τους μετανάστες, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι. Ε, χρειάζεται ε, ε, η κοινή πολιτική ασύλου θα αφαιρέσει την εθνική κυριαρχία ε, και θα έρχονται άνθρωποι χωρίς να δικαιούνται ε, άσυλο επειδή κινδυνεύουν. Ε, απλώς φτάνουν στις ακτές μας. Πρόκειται για μία περιορισμένη αντίδραση ισχνή απέναντι σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Αρνούμεθα να το αντιμετωπίσουμε και το μόνο που λέμε είναι είναι δύσκολο, ας αρχίσουμε να ανοιγόμαστε. όσοι μίλησαν με πάθος σήμερα υπέρ του ανοίγματο των συνόρων, ε, ίσως ε, ε, θα έπρεπε να δεχτούν να φιλοξενήσουν ορισμένους πρόσφυγες στα σπίτια τους. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, οι υπόλοιποι από εμάς θα τους παίρνανε πιο στα σοβαρά. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Άννα Ζαμπόρσκα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, Μιλούμε για την αρχή της δίκαιης αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών κατά την επίλυση ε, της προσφυγικής κρίσης. Ψήφισα υπέρ. Είμαι υπέρ όμως και της συνεπούς επιστροφής εκείνων των μεταναστών των οποίων η ζωή δεν απειλείται από την πείνα και τον πόλεμο. Βεβαίως ο καθένας έχει δικαίωμα για μια καλύτερη ζωή. Ε, η προτεραιότητα όμως δίνεται στη διάσωση των ανθρώπων που κινδυνεύουν. Ε, δεν μπόρεσα να υποστηρίξω στο, ε, την αύξηση των αριθμών πέραν των 40.000. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το Κοινοβούλιο όμως ε, θα πρέπει καταρχήν να περιμένει τη συμφωνία των κρατών μελών και μετά να αποφανθεί. Επίσης ε, δεν πιστεύω ότι από ένα προσωρινό μέτρο πρέπει να δημιουργηθεί ένας μακροπρόθεσμος διαρκής μηχανισμός και γι' αυτό στην τελική ψηφοφορία απήχα. Ο κύριος Ανδρέας Μαμίκινς επίσης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ υπερψήφισα αυτήν την ε, σοβαρή έκθεση και θα σας εξηγήσω γιατί. Το θέμα των προσφύγων ε, αφορά στην ουσία την ελληνική και τις ε, κοινέ αξίες και ντρέπομαι που συνάδελφοι από τη δική μου χώρα ε, που έρχονται από διαφορετικές πολιτικές ομάδες ε, την καταψήφισαν. Ε, δεν είναι δυνατόν εμείς να καθόμαστε εδώ μόνο για να καταναλώνουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 34 εκατομμύρια ευρώ έλαβε η χώρα μου για να βοηθήσει τους ε, ε, μετανάστες και θα λάβει ακόμα 29 εκατομμύρια επιπλέον. Ταυτόχρονα όμως λέμε και ότι δεν θέλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη για ανθρώπους που ε, ζουν δραματικές στιγμές στη ζωή τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανυψωθούμε και εμείς οι ίδιοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Μάριαν Χάρκιν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι διότι μπόρεσα να υποστηρίξω την έκθεση σήμερα που μιλάει για διανομή 40.000 προσφύγων σε άλλα κράτη-μέλη τα επόμενα δύο χρόνια, κυρίως από την Ελλάδα. Ε, αυτή ήταν μια ε, αντίδραση έκτακτης ανάγκης κατά παρέκκληση των υφισταμένων κανόνων. Μόνο οι ετούντες άσυλο που χρειάζονται όντως διεθνή προστασία θα είναι επιλέξιμοι. Ε, ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς είπε ότι αυτή είναι καθοριστική στιγμή στην ιστορία της Ευρώπης και ε, θα ήθελα ε, οι απλοί άνθρωποι να βοηθήσουν όσο μπορούν. Αυτό το κάνουν. Έχω δεχθεί πολλά emails από Ιρλανδούς που διαθέτουν βοήθεια. Τα σπίτια τους περηφανεύομαι που είμαι περήφανη που είμαι Ιρλανδή και Ευρωπαία όταν βλέπω τις επιτροπές που καλωσορίζουν τους πρόσφυγες. Επίσης, ο Πάπα είπε ότι κάθε ενορία θα πρέπει να ε, ε, φιλοξενήσει μια οικογένεια προσφύγων, τον άσυλο, ε, διότι αυτό βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε ε, τις δύο κατηγορίες ε, των προσφύγων. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα περαιτέρω βήμα καταργώντας το έθνος κράτος και την δυνατότητα των κυβερνήσεων να λαμβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις για θέματα τόσο σοβαρά όσο είναι η μετανάστευση και το άσυλο. Οι προτάσεις ε, ενώπιον του Κοινοβουλίου δεν αφορούν μόνο θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, έχουν την υπεροψία να αξιώνουν ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να αλλάξουμε και το διεθνές δίκαιο. Εμείς ε, επεκτείνουμε τον ορισμό του ασύλου και του πρόσφυγα για να συμπεριλάβουμε όλους τους φτωχού από όλες τις χώρες. Και έτσι λέμε στον κόσμο ότι ανοίγουμε τις πύλες μας στον καθένα από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία που δεν είναι ε, πραγματικός πρόσφυγας αλλά θέλει να ε, έρθει ως οικονομικός μετανάστης. Έτσι μειώνονται οι μισθοί ε, διαφορο... μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν φωνή στην Ευρώπη θα είναι αυτοί που δυνοπαθούν λόγω της αλαζονίας των ανθρώπων σε αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ συνάδελφε Βούλφ. Τέλος, τελευταία αιτιολόγηση, ο συνάδελφος Άρνοτ. Ε, ξεχάσαμε τη συλλογική μας μνήμη ε, υπάρχουν 25 ε, με 30 ε, πρόσφυγες στην Τουρκία ή Ορδανία που αντιστοιχούν σε ένα πρόσφυγα εδώ. Συχνά γίνεται το ταξίδι με την βοήθεια λαθρεμπόρων διακινητών. Ξεχνάμε την, ε, τα δεινά αυτών των ανθρώπων που μένουν πίσω. Να σκεφτούμε πριν δράσουμε. Η ανθρωπιστική κρίση δεν τελειώνει στα σύνορα της Ευρώπης. Ε, δεν θα πρέπει να ε, φερόμεθα έτσι προκαλώντας θανάτους που θέλουμε να παρεμποδίσουμε. Υπάρχουν έξι χώρες πλούσιες του κόλπου που δεν έχουν δεχθεί, υποδεχθεί ούτε έναν πρόσφυγα. Θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε και εκείνοι να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους. Ε, ο κόσμος ε, δεν τελειώνει στην Ευρώπη ε, και δεν θα πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία που χαρακτηρίζει την Ήπειρό Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε στην έκθεση αυτή για τα μέτρα Ιταλίας και, ε, για την Ιταλία και την Ελλάδα. Ε, η επόμενη έκθεση είναι η κυρία Κέρστιν Βέσφαλα, αστική διάσταση των πολιτικών. Θα είναι η τελευταία έκθεση ε, για την οποία θα επιτρέψουμε αιτιολογήσεις ψήφου. Είναι 7 οι συνάδελφοι, όμως είναι σχεδόν 3 παρατέταρτο και πρέπει να ετοιμαστεί η αίθουσα. η συνάδελφος Γκίλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 75% των ε, πολιτών της Ευρώπης, ε, δηλαδή 2 τρίτα του ΑΕΠ, ζουν σε αστικές περιοχές. Και αυτή είναι ακριβώς ε, η μεγάλη μας πρόκληση και μάλιστα και σε επίπεδο καθημερινότητας. Είναι εκεί που υποφέρουν οι άνθρωποι από την κλιματική αλλαγή, τον αποκλεισμό, την μόλυνση κτλ. Χρειάζεται λοιπόν καινοτομία. Πρέπει να αντιδράσουμε με καινούριε λύσεις. νομίζω ότι ε, στην δικιά μου χώρα και ειδικότερα στη δικιά μου περιοχή ε, έχουν γίνει πάρα πολλά. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει τα μάγιστα έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι περιοχές αυτές. Ωστόσο υπάρχει έλλειψη συντονισμού όσον αφορά την αστική πολιτική και οριζόντια αλλά και εγκάρσια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πόλεις μικρές και μεγάλες θα είναι πιο κοντά ε, στις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, και να εμπλακεί πλήρως ε, η, το, το αστικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με πολύ μεγάλη χαρά υποστήριξα την έκθεση αυτή, διότι μας είχε απασχολήσει το θέμα αυτό, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς ε, το σωστό βήμα να συζητήσουμε τα θέματα των πόλεων ή τη γεννητικότητα της πόλης. Ε, όντως έγινε πολύ καλή συζήτηση και όντως θα πρέπει να το συζητάει η Ευρώπη. Ε, είναι βεβαίως ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αστικό θεματολόγιο. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι Ευρωπαίοι που ζουν στις πόλεις και αυξάνεται και η μετακίνησή τους προς τις πόλεις, η αστιφιλία δηλαδή. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να στερείται τελείως ε, ε, αστικής πολιτικής. Δεν θα ήταν καλό αυτό και θα σήμαινε παρέτηση από τις μελλοντικές μας φιλοδοξίες. Πιστεύω ότι εκείνοι που καταψήφισαν την έκθεση αυτή θα το μετανιώσουν και ελπίζω να το ξανασκεφτούν διότι η κινητικότητα στις πόλεις είναι αστική, και η αστική πολιτική είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Ευχαριστώ κύριε Πόλτσακ, η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άμεσο ε, αντίκτυπο στις ε, ε, εθνικές πολιτικές για, την, για τις αστικές περιοχές. Θέλουμε πολιτική η οποία να είναι βιώσιμη, η οποία να είναι ανεκτική και η οποία να είναι πράσινη και καινοτόμα. Οι φιλοδοξίες είναι μεγάλες και οπωσδήποτε θα πρέπει να βελτιωθεί η αστική διάσταση των πολιτικών της Ευρώπης και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της απλούστευσης της ε, διαδικασίας ε, ε, απόδοση των κονδυλίων και καταμερισμού των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αστικές περιφέρειες είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι πολυπληθείς. Πρέπει να γίνουν και λειτουργικές και επομένως οι περιφέρειες, οι πόλεις, οι τοπικές αρχές, οι εθνικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστούν αλλά να ακούν και την γνώμη των ντόπιων γιατί αυτοί ξέρουν ποιες είναι ε, κυρίαρχα οι ανάγκες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακοβέη. Ο κύριος Μπάλτσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο. Εγώ θεωρώ θεμητό να συζητάει το Κοινοβούλιο έκθεση που αφορά την αστική διάσταση της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι λογικό γιατί το 80% των πολιτών της Ένωσης ζει στις πόλεις. Αλλά δεν είναι θετική η εξέλιξη αυτή. Δυστυχώς σε πολλές χώρες ε, ο κόσμος εγκαταλείπει την Ήπεθρο γιατί η κατάσταση είναι αβίωτη, διότι έχει ρημάξει η γεωργία, έχει γίνει βιομηχανική παραγωγή και είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας αυτό και στις περιφερειακές πολιτικές και να το συζητούμε. Τι θέλουμε να κάνουμε στην πόλη. Γιατί λοιπόν ψήφισα αποχή εγώ. Διότι υπήρχε μία παράγραφος μέσα στην έκθεση που λέγει ότι αποσκοπούν στην ίδρυση ενός κεντρικού θεσμικού οργάνου ε, δίπλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή τη συγκέντρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπάλτσο. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Υποστήριξα την έκθεση για την αστική διάσταση των πολιτικών της Ένωσης. Πολλές ενώσεις, σύλλογοι ασχολούνται με την αστική πολιτική, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ακούσαμε ήδη ότι 50 με 80% του πληθυσμού στις μεγαλού ζει στις μεγαλοπόλεις και αυτό συνεπάγεται πολλά καθημερινά προβλήματα. Ε, υπάρχουν περιβαλλοντικές επιρροές, ε, υπάρχουν διακινούμενοι εργαζόμενοι. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και να λυθούν ως τα προβλήματα αυτά. Ε, επίσης θα πρέπει να δούμε τη συνύπαρξη πόλης με το περιβάλλον της. Δηλαδή οι αστικές κοντινές μεταφορές πρέπει να ενισχυθούν και θα πρέπει να ανταλλάσσουμε παραδείγματα καλής πρακτικής στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι το πλέον ενδεδειγμένο για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ ε, ο συνάδελφος Κέλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με χαρά υποστήριξα την έκθεση, ψήφισα με την ομάδα μου σε όλες αυτές τις ψηφοφορίες ήταν ενδιαφέρον και ικανοποιητικό ότι σημείωσα ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο ήταν υπέρ. Δεν εκπλήσει αυτό αφού ο μισός πληθυσμός της γης ζει σε αστικές περιοχές, το 75% ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τις πόλεις μας, τις μεγαλοπόλεις μας, να τις αναβαθμίσουμε ε, προάγοντας και την οικονομική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση, ο αθλητισμός πρέπει να παρέχονται στους νέους θέσεις εργασίας για τους ενήλικες και μια καλή ζωή για όλους. Και η καθαρή ατμόσφαιρα θα πρέπει να διασφαλίζεται στις πόλεις. Για να γίνει αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις μεταφορές, περισσότερα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα, ποδήλατα, ε, δηλαδή οχήματα που δεν έχουν μεγάλα, πολλές εκπομπές. Πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Κέλλη. Ο συνάδελφος Μαμίκινης. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Παράλληλα όμως Νομίζω ότι αυτή είναι μια επίκαιρη απόφαση. Ε, αναφέρθηκε ότι πάνω από 75% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε αστικές περιοχές. Ε, μεγάλες και οι μεγάλες πόλεις, οι μεσαίες, μικρές πόλεις είναι πολύ σημαντικές ε, και για τον πολιτισμό και για τη βιομηχανία. Ε, οι ε, αυτές οι νηστώσεις συνενώνονται και αυτό παρουσιάζεται και ανάγλυφα στις πόλεις μας εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Θα πρέπει η αστική διάσταση να συντονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό δεσμευτικό σήμερα, αλλά είναι σημαντικό θέμα. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε δηλαδή κοινή στρατηγική και για να ε, την εφαρμόσουμε θα πρέπει να εντάξουμε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στο έργο μας. Υπάρχει κάποιο κενό μεταξύ ε, δήμων και εθνικών κυβερνήσεων και θα πρέπει να τονίσω πάλι ότι ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάμικίνσε και τέλος ο συνάδελφος Έθεριτζ. Ευχαριστώ. Οι ανοιχτέ πολιτικέ της Ένωση είναι προσπάθεια παράκαμψης του έθνους κράτους ώστε οι ευρωπαϊκές πολιτικές να δικαταστήσουν τις ε, ε, πολιτικές της περιφέρειας. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να προειδοποιήσουμε ότι αν συμβεί αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για θετικές διακρίσεις όταν πρόκειται για απασχολουμένους στα δημοτικά συμβούλια. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να καταβάλλετε ένα τίμημα ε, μετά από την πολιτική αυτή ε, ε, γιατί οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε σε τοπικό επίπεδο τα κονδύλια εκεί όπου χρειάζεται. Εάν παρεμβαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι αντιδημοκρατικό και απομακρύνουμε τη δημοκρατία από το επίπεδο του λαού. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ιδέα αυτή και να ε, αποτρέψουμε την ε, εξάπλωσή της ε, και την εφαρμογή της. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκαν οι αιτιολογίες ψήφου για την έκθεση Βέστφαλ.